Ας αρχίσουμε κυρίες και κύριοι, λέει ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Παρακαλώ καθίστε. Δεκάτησα θεωρή διακόπη συνεδρίαση και την την συνέχεια και έχουμε εγκρίνει διάφορα έγγραφα σε σχέση με αυτά τα οποία φέσαμε τότε. Έχετε λάβει τα έγγραφα, δεν βλέπω καμία ένσταση, επομένω ε, τα πρακτικά των σχετικών συνεδριάσεων